Έλαβα επίση από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ετήματα για ορισμό σε επιτρέπες και αντιπροσωπείες. Ε, Βρίσκονται στα πρακτικά τη σημερινή συνεδρίασης. Εάν δεν υπάρξει καμία παρατήρηση από εδώ μέχρι την έγκριση ε, των πρακτικών, θα θεωρήσουμε ότι